zmiana regulaminu pracowniczego urzędników wspólnot europejskich i warunków zatrudnienia. Έχουμε επίση την έκθεση του κυρίου Ράπκαη για την, ε, τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώ και του καθεστώτο που εφαρμόζεται στο ελληνικό προσωπικό των κοινοτήτων αυτών. Επίση έχουμε τι εκθέσει Γκουαλτιέρη και Σουριάν σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού για το τμήμα υπαριθμών 2, το τμήμα 3 και το τμήμα 10. Το φορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπατε εκπρόσωπε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε και κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, οι οποίοι βρίσκονται καθοδόν, έχουν μείνει μάλλον στην κυκλοφοριακή κίνηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώνουμε το τελικό βήμα μιας συναρπαστικής νομοθετικής και διοργανικής περιπέτειας τετραμερούς διαλόγου, δηλαδή την θέσπιση μιας αποτελεσματικής, φιλόδοξης και στραμμένης προς το μέλλον Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης το κείμενο που έχουμε με τροποποίηση του κανονισμού προσωπικού, του νοσονομικού κανονισμού και τον διορθωτικό προπολογισμό που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα και θα ψηφίσουμε αύριο, αποτελούν την ε, έκβαση, επιτυχή έκβαση μηνών διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Όλων ενωμένων σε ένα κοινό στόχο, το πώς δηλαδή θα οργανωθεί ο τρόπος με τον οποίο ακούγεται η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα εισακούεται αυτή η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Εμείς από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλη σοβαρότητα τις ευθύνε μας στην περιπέτεια αυτή, στη διαπραγμάτευση αυτή με κύριο γνώμονα την, στη δράση αυτή τη υπηρεσία εξωτερική δράσεω την επικράτηση του κοινοτικού συμφέροντος, του κοινού συμφέροντος. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν θα ξεχθεί σήμερα η συζήτηση και έτσι περαιτέρω με αυτό το πνεύμα προσμένουμε με δημονία την, θέση σε, την επίσημη θέση σε λειτουργία τη υπηρεσία εξωτερική δράσης το Δεκέμβριο του 2010 μόλι ένα χρόνο μετά τη θέση εφαρμογή της συνθήκης, θέση ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα. Ξεκινάμε ακούγοντα πρώτα του εισηγητές μα, Η κυρία Γκρέσλιν η πρώτη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε Σεύσκοβης, κύριε Επίτροπε Λεβαντόφσκη, κυρία Αντιπρόεδρε, ε, αν είπατε εκπρόσωποι, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να πω ότι δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσει την ανάληψη δράσεως αυτή η υπηρεσία, η ΕΕΔ, μέχρι να δούμε τα, τα αποτελέσματα της δράσης της. Έχουμε δει από την ε, εμπειρία μας ότι είναι όρος εκ κάφων νεφ για την ε, αποτελεσματική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο συνέπραξε στη θέσπιση της. Πρόκειται για μια τέρα incognita, ένα νέο δηλαδή πεδίο δράσης, όπου ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλες προκλήσεις και ως αρμόδια για τα θέματα του ελέγχου του προϋπολογισμού παραμένω πάντοτε σε επαγρύπνηση ως προς την αποτελεσματικότητα αλλά και την δυνατότητα ελέγχου των δημοσιονομικών αυτής τη υπηρεσία, Είναι μαζί με τη, στην κοινή μα έκθεση μα με τον κύριο Ριβελίνη αυτό το μέλημα το οποίο έχουμε προβάλλει προσπαθώντα να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ε, ορίζοντας τους υπεύθυνους και του τους υπόχρεους προς λογοδοσία, ορίζοντας ως κύρια αρχή και υποχρεωτική την ε, διαφάνεια, την υποχρέωση για λογοδοσία και καθιστώντας ξεκάθαρο ότι πρέπει να έχουν οι ελεκτικές αρχές το ρόλο κλειδί στην υπόθεση αυτή. Έχουμε προσδιορίσει μέσα από την έκθεση δυνατότητες και διατάξεις περί συνεργασίας, σύμπραξης των υπηρεσιών που μπορούν να ή οφείλουν να ελέγχουν τη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο και η ασωμάτωσή του στον προπολογισμό παραμένει ένα θέμα επικαιρότητα, όπω ακριβώ και η απαλλαγή του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ όλους για την ε, συνεργασία που επέτρεψε την θέσπιση αυτής της ε, αυτής της εκθέσεως, τους συνεργάτες με τους οποίους συντάξαμε την Επιτροπή και ιδιαίτερα τη Βελγική Προεδρία η οποία μας, ε, μας συνέδραμε πολύ στην υπόθεση αυτή. Θέλουμε λοιπόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που δεν είναι δεδομένη μόνο με την συγχώνευση των υπηρεσιών. Το 10% το λαμβάνει λοιπόν η ΕΕΔ. Κύριε Πρόεδρε, έχω τρία λεπτά. Ο Πρόεδρος διέκοψε την ομιλήτρια. Είπαμε να σας δώσουμε δύο λεπτά τώρα και ένα στο τέλος, λέει ο Πρόεδρος. Αν προτιμάτε, μπορείτε να εξατλήσετε και τα τρία σας λεπτά τώρα. Καλώς, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μια υπηρεσία λοιπόν η οποία είναι επαγγελματική μόνο εφόσον μπορεί να γνωρίζει ξεκάθαρα τα καθήκοντα τα οποία έχει επομιστεί και γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε να αναλάβει δράση και να επανέλθουμε το χύτερο δυνατό στην επανεξέταση αυτών των δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη σημασία λοιπόν έχει η ανάπτυξη των διπλωματικών δράσεων Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάπτυξη δράσης εξωτερικής ε, στις ε, χώρες του υπόλοιπου κόσμου κατά τρόπο ώστε να ξαναδιατυπωθεί ο, χάρτη χάρτης της διπλωματίας ανά τον κόσμο είναι πιστεύω η υπηρεσία εξωτερικής δράσης αυτό που χρειαζόμαστε για να εκπροσωπήσει την Ευρώπη σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Um, ώρα σας, ε, τρία λεπτά. Φεστένσιο Ριβελίνη, έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, λέει Ο δημοσιονομικός κανονισμός για την ΕΕΔ και για τις αρχές και τους κανόνες βάσης που θα ορίζουν τον προϋπολογισμό της νέας διπλωματικής υπηρεσίας που δημιουργήθηκε από τη συνθήκη της Λισαβόνας και που θα ρυθμίζει το υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων που θα αντιπροσωπεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξωτερική πολιτική είναι κάτι το εξαιρετικό. Η υπηρεσία έτσι όπως διαρθρώθηκε ενίχευε διάφορους κινδύνους και αυτό λόγω της αποκεντρωμένης της φύσης με σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή η ευθύνη των διαχειριστών που θα έπρεπε να διαχειριστούν εκατοντάδες ε, εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να οδηγήσει σε απάτες και καταχρήσει σε βάρος ε, του κοινοτικού προϋπολογισμού. Υπάρχει, υπάρχουν εξουσίες ε, του Κοινοβουλίου το οποίο ως εκπρόσωπος των Ευρωπαίων πολιτών θα έπρεπε να έχει λόγο αλλά ο αρχικός διάλογος έγινε μεταξύ Κομισιών και Συμβουλίου που θέλησαν να διαρθρώσουν αυτήν την υπηρεσία με διακυβερνητική λογική και κατά της κοινοτικής μεθόδου. Μετά από διαπραγματεύσεις με τη Βελγική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταλήξαμε σε μια συμφωνία που ενίσχυσε το ρόλο του Κοινοβουλίου και το κατέστησε δικαιούχο στη συζήτηση. Βασικά σημεία τώρα. Η Κομισιόν θα υποβάλει στο σχέδιο προϋπολογισμού ως παράρτημα μία αναλυτική πρόταση όπου θα έχουμε όλα τα διοικητικά και λειτουργικά έξοδα της ΕΕΔ και όπου θα συμπεριλαμβάνεται και η ΚΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Το άρθρο 1 στο οποίο αναφέρονται όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα δίνεται η υποχρέωση στο Διευθυντή να υποβάλει τη σχετική αναλυτική έκθεση κάθε χρόνο προς ε, το Κοινοβούλιο. Ζητάμε επίσης να υπάρχει ένας κοινός λογιστής ο οποίος θα ελέγχει τους λογαριασμούς με μία ρήτρα αναθεώρηση το 2013. Επίσης γίνεται αναφορά και στο εποχιακό προσωπικό. Υπάρχουν όμως ακόμη θέματα προς συζήτηση, τα οποία θα συζητηθούν στην τριετή αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Και το θέμα που εκκρεμεί λοιπόν είναι η απαλλαγή του οργάνου και η διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μέσα στα πλαίσια του Γενικού Προϋπολογισμού. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση για το Κοινοβούλιο. Αξιολογήθηκε ο κεντρικός του ρόλος συμπεριλήφθηκαν στη συζήτηση όλα τα όργανα. Ο χρόνος σας λέει ο Πρόεδρος. Το γεγονός ότι έχουμε έναν κοινό λογιστή ελεγκτή για τα όργανα είναι μια πολύ καλή δουλειά του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίση, εξαιρετήσατε το χρόνο σα. Ο κύριο Ράπκα έχει το λόγο. Έχει συνολικά 6 λεπτά. 4 συν 2. Να σα προτείνω να το κάνουμε 4 συν 2. 4 τώρα και 2 στο τέλο. Βεβαίω, Πρόεδρε. Ας δούμε όμως πόσα θα χρειαστώ τώρα και αν περισσέψει κάτι στο τέλος ε, για να απαντήσω στι αντιδράσει. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Έστον, όταν, ε, κυρία Εσεύκοβιτς, όταν λέω αγαπητοί συνάδελφοι, εννοώ και εσάς όπως και τους εκπροσώπους της Προεδρίας Συμβουλίου. Και αυτό γιατί η δουλειά μας ήταν πράγματι συνεργατική. Χωρίς αυτή τη συνεργασία δεν είχαμε καταλήξει στο αποτέλεσμα το οποίο έχουμε σήμερα να συστήσουμε. Είμαι τόσο ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στο το κομμάτι το οποίο ε, απασχόλησε εμένα και στο οποίο είχα την επιτήρηση, την εποπτεία. Και θέλω να πω ότι Ήτανε, Πρόεδρε, πολύ καλή ιδέα που είχατε εγκαίρως ήδη με την έκθεση Μπροκ Φερχόφστατ Κουαλτιέρη να προσκαλέσετε σε μια κοινή ανταλλαγή απόψεων όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Διότι έτσι ήταν ξεκάθαρο για αυτούς που αναλάμβαναν το έργο που παρέδιδαν η προηγούμενη η προηγούμενη ομάδα, ότι έχει γίνει κάποια προκαταρκτική εργασία και πάνω σε αυτή θα πρέπει να στηριχθούν. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την θέση σε λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσεως. Ε, καθαρά οργανωτικά θα τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός προσωπικού εκεί όπου χρειάζεται να εφαρμοστεί αυτός. Οργανωτικά, είπα. Η οργάνωση όμως είναι πολιτική και η πολιτική είναι επίσης οργάνωση. Και άρα στις διαπραγματεύσεις το είδαμε αυτό όταν ασχοληθήκαμε δηλαδή με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης ότι χωρούσε κάποια διαφορετική ενδεχομένως ερμηνεία από αυτήν στην οποία καταλήγαμε. Πρόβλημα όμως και δίλημα το οποίο τελικά επιλύσαμε σε αγαστό κλίμα συνεργασίας. Τι θέλαμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε με τον κανονισμό προσωπικού. Θέλαμε οι τρεις συνιστώσεις, όπως αναφέρθηκαν νωρίτερα, του προσωπικού να έχουν ισότιμη μεταχείριση. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με προσωπικό που θα ε, αποσπαστεί από την Επιτροπή, άλλο που προέρχεται από το Συμβούλιο και άλλη μια κατηγορία προσωπικού από τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Εκεί ακριβώς είχαμε το πιο δύσκολο σημείο, γιατί ήταν καινοφανές το έχουμε προσωπικό από τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών και εκεί είπαμε ότι θα υπάρχει μια προσέγγιση όπου θα ξεχωρίζουμε την κοινοτική ε, απασχόληση ή ε, ανάθεση και την εθνική ανάθεση. Προτείναμε λοιπόν την κοινοτική προσέγγιση, στην οποία νομίζω μπορούμε να δούμε τα περισσότερα πλέον εκτήματα και να είμαστε ικανοποιημένοι. Ταυτόχρονα είπαμε ότι θέλουμε ισορροπημένη εκπροσώπηση των δύο φύλων και γεωγραφική εκπροσώπηση ισορροπημένη. Ιδιαίτερα λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ως προς τη διάσταση της ισότητας των δύο φίλων και κυρία Άστον πρέπει να πω ότι και εσείς επιπλέον των όσων είχαμε δεσμευτικά ορίσει μέσα στη συνθήκη κάνατε δηλώσεις οι οποίες ακριβώς αποτελούν ε, αναπόσπαστο τμήμα πλέον αυτού του πακέτου συμφωνίας και έτσι και οι δύο διαστάσεις ισότιμης μεταχείρισης του φύλου δηλαδή και της γεωγραφικής προέλευσης ή καταγωγής είναι πιστεύω εδρεωμένες μέσα στην ε, στις αρχές που διέπουν το προσωπικό αυτής της υπηρεσίας. Ταυτόχρονα έχουμε και την αρχή της πίστης. Πίστη προς την υπηρεσία, προς τον την είπα το εκπρόσωπο, το δικαίωμα άρνηση κυρίας από τις διπλωματικές υπηρεσίες με δυνατότητα ενδεχόμενης παράτασης τους απασχόλησης των ε, υπαλλήλων που προχωρούν από τι διπλωματικές υπηρεσίε. Ήταν μια σειρά από προβλήματα που μπορούσαμε να λύσουμε και κάτι ακόμη που δεν θα πρέπει να ε, το οποίο δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε τη σημασία. Η νέα αυτή διπλωματική υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Διπλωματική Υπηρεσία, χρειάζεται ταυτότητα. Θέλετε, χρειάζεται ίδια ταυτότητα. Κάτι το οποίο δεν προβλεπόταν από τι συνθήκε. Χρειάζεται δηλαδή να γνωρίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί ότι έχουν τη δυνατότητα για μια κοινή και περαιτέρω κατάρτιση, μετεκπαίδευση Και ήθελα να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι δεν ήταν αυτονόητο από τον κανονισμό ότι θα προβλεπόταν αυτή η δυνατότητα, αλλά γι' αυτό και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστώ την υπατή εκπρόσωπο, διότι μας είπε, μας εξήγησε, δήλωσε ξεκάθαρα πόσο σημαντική θεωρεί αυτή τη δυνατότητα και γι' αυτό την καλύπτει μέσα από την δήλωσή της, δήλωση η οποία δεν αποτελεί έγγραφο ισοδύναμο ίσως με τον κανονισμό του προσωπικού, ε, δεν ανήκει, δεν είναι άρθρο του κανονισμού του προσωπικού, αλλά πάντως καθησυχάζει όλους εμάς που θα θέλαμε να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Και έτσι από την 1η Δεκεμβρίου μπορεί πια να ανοίξει τα φτερά της αυτή η υπηρεσία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Έχετε ακόμη ένα λεπτό για το τέλος της συζήτησης. τώρα δίνω τον λόγο στον συνάδελφο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Άστον, κύριε Επίτροπη. Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέσπιση ενός νέου, νέου τμήματος του προϋπολογισμού για την ΕΕΔ και τις πρόσθετες δαπάνες για το προσωπικό. Αυτό εκφράζει τη βούληση για τη γέννηση αυτής της νέας υπηρεσίας που χρειάζεται η Ευρώπη και είναι κατεπήγον. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει η αρχή του προϋπολογισμού να μην συζητήσει όλες τις πτυχές του προϋπολογισμού για τη διαχείριση του οργάνου και του προσωπικού του. Οι κανονισμοί που θα εγκρίνουμε ενισχύουν τα αποτελέσματα της Συμφωνίας της Μαδρίτης και προχωρούν και πιο πέρα. Και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Γκρέσλερ, Ράπκα, Ιβελίνη όπως επίσης και την κυρία Άστον και τον Πολ Κριστόφερσον. Ο κανονισμός εγγυάται ότι όλοι οι υπαλλήλοι της υπηρεσίας θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις ασχέτως από πού προέρχονται. Και επίσης ζητείται να εγγυηθούμε την εθνική εκπροσώπηση, τη γεωγραφική εκπροσώπηση και το φύλλο. Αυτό αποφεύγει όμως, το Κοινοβούλιο όμως απέφυγε να θεσπίσει ποσοστώσεις οι οποίες θα ήταν λανθασμένες Επίσης θεσπίζονται έλεγχοι και ενισχύεται ο ρόλος της Κομισιόν. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε επιτυχία στις ειδικέ γραμμές του προϋπολογισμού για την ΕΕΔ ε, που επιτρέπουν το Κοινοβούλιο να ασκήσει περαιτέρω έλεγχο στην ΚΕΠΑ. Θα έχουμε μία εξωτερική υπηρεσία δράσης πιο ισχυρή, πιο κοινοτική, η οποία θα υπόκειται σε έναν γενικότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο αυστηρό και απαιτητικό, με ευθύνη και με επικοδομητικό πνεύμα, με στόχο να βοηθήσουμε τον ύπατο εκπρόσωπο σε αυτήν την τιτάνικη την τιτανική προσπάθεια, τιτάνια προσπάθεια να ενισχύσει την Ευρώπη με μια διπλωματική υπηρεσία. Έχετε ακόμη ένα λεπτό στο τέλος της συζήτησής μας. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος Λάσλο Σούριαν. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με χαρά σημειώνω ότι έχουμε εδώ παρόντες και το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια συνεδρίαση όπου συζητούσαμε τον δημοσιονομικό σχεδιασμό το 2010 και μετά. Είχαμε πει σε τι είδους πόρους μπορούμε να στηρίξουμε αυτήν την ε, ε, λειτουργεί αυτή τη υπηρεσία. Μα είχε απαντήσει τότε η Επιτροπή, δεν χρειάζεται θα κάνουμε απλώ μεταφορέ ε, κονδυλίων. Όμω δεν είχαμε συμφωνήσει, δεν είχαμε πιστεί και τα όντι έγιναν κάποιε μεταφορέ κονδυλίων που κάλυψαν κάποιε ανάγκε, όμω χρειάστηκε συνολικά να, διατεθούν, να εξευρεθούν 44 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για επιπλέον δαπάνε που καλύπτουν τις ανάγκες για ένα τρίμηνο. Και πρέπει να κατανεμηθούν ισότιμα. Ακόμη δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, έχει μόνο το 10% του, του προσωπικού της και πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το ποσό αυτό το οποίο θα εγκρίνουμε αύριο θα χρειαστεί να διαρκέσει να χρηματοδοτήσει δράσεις που θα κρατήσουν περισσότερο διάστημα από ό,τι αρχικά έχει προβλεφθεί. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να είχαμε προβλέψει περισσότερο επιπλέον κονδύλια. Εν πάση περιπτώσει όμως θεωρώ ότι είναι καλό το να μπορεί το Συμβούλιο τώρα να ε, δείχνει μια γενεοδορία στην υπόθεση αυτή ώστε να υπάρξει και η αναγκαία ορατότητα για, το, ε, για την κοινή γνώμη του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η συνθήκη της, αγώ, της Λεσσαβόνας. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως υπόθηκε νωρίτερα, έχουμε δώσει στην αναλογική εκπροσώπηση, τη γεωγραφική κατανομή και προσπαθήσαμε να είμαστε στο δυνατόν πιο ευέλικτοι για να μπορέσει ταχύτατα να αναλάβει δράση η υπηρεσία. Ελπίζουμε από εδώ και μπρο ότι τα ποσά που θα εγκριθούν θα αξιοποιηθούν κατά τρόπο φιδωλό, κατά τρόπο οικονομικό και αποτελεσματικό και κλείνοντα θα ήθελα να πω ότι προσβλέπουμε σε μια πολύ στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη συμπληρωματική δράση την οποία, ε, η οποία πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πολλά ε, πόρων ε, πολλά από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή θα δούνε ότι χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξοικονομούν χρήματα. Πρόεδρε, Ελπίζω αύριο να εγκριθεί το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι για τις παρατηρήσεις σου και τώρα θα ήθελα for the και τώρα Α, ζητάτε το λόγο. Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Θα διακόψω τη συζήτηση για να ενημερώσω ότι εισέβαλαν στο Τσετσενικό Κοινοβούλιο σήμερα το βράδυ τρεις τρομοκράτες, κράτησαν ομήρους, προσωπικό, ε, βουλευτές και πρέπει να καταδικάσει το Κοινοβούλιο μας τέτοιου είδους τρομοκρατικές ε, δράσεις, να εκφράσει την ε, υποστήριξή του και τα συλληπιτήριά του στα θύματα της οικογένειας των θυμάτων, και νομίζω ότι ή δυνατόν θα ήταν καλό να ε, εισαχθεί ένα θέμα σχετικό με το Βόρειο Κάφκασο στην ημερή συντάταξη ακόμη για αυτή την εβδομάδα και συζητώ συγγνώμη για άλλη μια φορά που διέκοψα τις συζητήσεις. Ναι, ευχαριστώ για αυτές τις πληροφορίες και τις ειδήσει. Βεβαίως, εμείς καταδικάζουμε κάθε πράξη τρομοκρατίας και σε αυτή την περίπτωση είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η πράξη διότι ε, ήταν κατά του Κοινοβουλίου, επίθεση κατά του Κοινοβουλίου και εκφράζουμε την συμπάθειά μας ε, σε αυτούς που επλήγησαν. Ε, θα δοθεί επίσημα η είδηση αυτή αργότερα. Ευχαριστώ πολύ που επισήρατε την προσοχή μας πάνω σε αυτό το συμβάν. Ο επόμενος ομιλητής, ο Αντιπρόεδρος Μάρος Σεφτσοβίτς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ευχαριστήσω τον κύριο ε, Πλάκας που ε, μας ε, έδωσε αυτή την είδηση και εμείς η Επιτροπή καταδικάζουμε αυτή την πράξη και θα δράσουμε κατά συνέπεια. Θα ήθελα να επανέλθουμε στη συζήτησή μας και θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τον ε, εισηγητή κύριο Ραπκά για την εξαίρετη εργασία του ε, σχετικά με την πρόταση προς το Κοινοβούλιο. Είχαμε μια αγαστή συνεργασία τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες για αυτό το δύσκολο θέμα. Επίσης συγχαίρω τους κοιόδης εισηγητέ και επίσης ε, τις Επιτροπές Γιουρ και ΑΦΕΤ που εργάστηκαν κοπιοδός κατά τη διάρκεια όλες τις διαδικασίες. Επίσης εκφράζω την Τη της για την σκληρή εργασία που θα επιτρέψει ε, να ε, λειτουργήσει καλά ε, η ΕΔ σε σύντομο χρονικό διάστημα ε, ότι θα έχουμε τα θεμέλια, τα διοικητικά, τα οικονομικά για την υπηρεσία που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την λειτουργία της υπηρεσίας. Ε, συμμετείχα στη συζήτηση για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, και στη Μαδρίτη στον τετραμερή διάλογο εκπροσώπησα την Επιτροπή. Είναι σημαντική η συμβολή των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπροκ, Γκουαλτιέρη που συμμετείχαν στα αποτελέσματα της συζήτησης για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι η συμβολή τους στη συζήτηση ήταν σημαντική, ούτω ώστε η υπηρεσία αυτή να γίνει ε, μια ε, πραγματικά αποτελεσματική διπλωματική υπηρεσία. Αυτό ισχύει και για τον κύριο Ραπκάη, τον εισηγητή σα. Η τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων φαίνεται ότι είναι διοικητική, αλλά δεν είναι. Θα επιτρέψει την καλή λειτουργία ε, τη υπηρεσία προστασίας προς το ευρωπαϊκό συμφέρον. Βεβαίως είναι καλό το αποτέλεσμα του κυρίου Ραπκάη, η τροποποίηση και νομίζω ότι οι τροπολογίες βελτιώνουν το όλο κείμενο και θα ήθελα να αναφέρω μερικά βασικά στοιχεία της πρότασης. Όπως γνωρίζετε στην αρχική φάση θα έχει ε, τα τρία, ε, την Επιτροπή, το Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και τους εθνικούς διπλωμάτες ε, και το τμήμα θα μεταφερθεί το αρμόδιο του Συμβουλίου και της Επιτροπής στην υπηρεσία ε, και θα έχουμε το, τους υπαλλήλους θα, ε, και θα έχουμε τις κενές θέσεις που πρέπει να πληρωθούν. Από την 1η Ιουλίου ε, έχουμε ε, αξιωματούχους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα μπορέσουν ε, να ε, έχουν ίση μεταχείριση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις στην υπηρεσία και θα έχουμε τις προβλέψεις για το προσωπικό που θα εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την συμφωνία με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέκα χρόνια επιπλέον ε, τα κράτη θα παρέχουν διπλωμάτες ε, που θα εργαστούν στην υπηρεσία. Ο συμβιβασμός επίσης περιλαμβάνει ε, διευθετήσεις για να έχουμε μια ισορροπία γεωγραφική και ισορροπία ως προς το φύλλο. Ε, θα αναθεωρήσουμε την κατάσταση το 2013 και θα παρουσιαστεί μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Ξέρω ότι μερικοί από εσά εδώ θα ήθελαν ε, διευθετήσεις πολύ ισχυρότερο ενώ άλλοι είναι αντίθετοι. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι οι τροπολογίες που έχετε τώρα αποτελούν μια ισορροπημένη λύση. Οι διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό δεν ήσαν πάντοτε εύκολες. Η προπερασκευαστική εργασία ήταν περίπλοκη διότι χρειάζονται διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους του προσωπικού αλλά οι εργόδεις ε, προσπάθειες απέδωσαν πολύ καλά αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις. Έχετε αυτή την καλή πρόταση ενώπιόν σας και ελπίζω ότι αύριο οι τροπολογίες αυτές θα υιοθετηθούν από το Κοινοβούλιο και θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή είναι δεσμευμένη ούτω ώστε να υπάρξει μια καλή υπηρεσία εξωτερικής δράσης και ε, θα παρέχει κάθε βοήθεια σε αυτή τη νέα υπηρεσία. Ελπίζω ότι αύριο ε, θα είναι ιστορική ημέρα η οποία θα οδηγήσει στην ε, δημιουργία και ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και στην καλή λειτουργία της. Επόμενος ομιλητής, ο Γιάννους Λεβαντόφσκι. Κύριε, σας δίνω τον λόγο κύριε Πίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, αυτό το οποίο συζητούμε σήμερα είναι μια καλή απαρχή μιας μακράς ημέρας σχετικά με τον προϋπολογισμό. Βεβαίως, η εκκίνηση της, ε, εξωτερικής, ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής χρειάζεται ε, προϋπολογισμό και κανονισμό αλλά ε, αλλά ακολουθώντας ε, αυτήν την ε, διαδικασία, γι' αυτό τροποποιούμε τον κανονισμό υπηρεσιακή κατάστασης. Χαίρομαι που θα μπορούμε, που μπορέσαμε την περασμένη εβδομάδα στον τριμερή διάλογο να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα βάσει της συνθήκης της Λισαβόνα, ούτω ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ε, στην υπηρεσία εξωτερική δράση μια βάση στέρεα και αποδοτική. Βεβαίω, Έχουμε ασχοληθεί με πολλές ε, λεπτομέρειες ε, και για να μπορέσουμε να έχουμε ένα τμήμα του προϋπολογισμού για τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών και θα μπορέσει αυτό το τμήμα του προϋπολογισμού ε, να έχει έναν υπόλογο της Επιτροπής και να έχει έλεγχο επίσης. Ευχαριστώ λοιπόν τους εισηγητές ε, Γκρέσλερ, Ριβελίνη για την επικοδομητική ε, προσέγγιση. Επίσης έχουμε τον, ε, τροποποίηση του τμήματος 6 και η αρχή επί του προϋπολογισμού νομίζω ότι θα μπορέσει τώρα να εγκρίνει τον τροποποιητικό ε, ε, προϋπολογισμό ε, χωρίς τροπολογία ούτω ώστε να μπορέσει να αρχίσει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Η πρώτη δόση θα μπορέσει να καλύψει μέχρι το 2013 τις δραστηριότητες και αυτή είναι η δέσμευσή μας να έχουμε το 1 τρίτο του προσωπικού να προέρχεται από το διπλωματικό σώμα των κρατών μελών. Τούτων λεχθέντων καλό το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει τον τροποποιητικό διορθωτικό προϋπολογισμό ε, του Συμβουλίου και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου ε, και επίση ε, στον κύριο Σούριαν και Γκουαλτιέρη, τους εισηγητές. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις παρατηρήσεις σας. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, είπα το εκπρόσωπο, Lady Ashton περιμένουμε ε, την παρέμβασή σας. Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριε και κύριοι βουλευτές, λαμβάνω το λόγο πολύ σύντομα, μόνο και μόνο για να ευχαριστώ τους συζητητές, κυρία Γκρέσλε, τον κύριο Κουαλτσέρη, τον κύριο Ραπκάη, Χάρη στη δική τους δουλειά και τη συνεργασία των βουλευτών ε, του Κοινοβουλίου μπορέσαμε να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Ξέρω ότι ήταν ε, μερικές φορές σκληρές οι διαπραγματεύσεις και ήσασταν σκληροί διαπραγματευτές. Όμως το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα να συζητήσουμε είναι καλό αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα το οποίο αντικατοπτρίζει στην ουσία το πνεύμα της συνθήκης Λισαβόνας κατά την εφαρμογή της με σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον. Ήταν, όπω είπα, σκληρή δουλειά. Ευχαριστώ όλους σας για τη δουλειά αυτή και πιστεύω ότι πάνω απ' όλα ρίχνουμε τα θεμέλια μιας τέτοια υπηρεσία που θα ε, επιτρέψει την εμπλοκή του Κοινοβουλίου στο μέλλον στις εργασίες της και εγώ προσωπικώς έχω δεσμευθεί για απόλυτη διαφάνεια. Επίσης, πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία θα πρέπει να εκφράζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να την αντικατοπτρίζει εις βάθος και εις ύψος και εις πλάτος. Ε, κάθε κράτος μέλος, κάθε εκπρόσωπος ε, κράτους μέλους επιτροπής θα πρέπει να αισθάνονται υπερηφάνεια και να βλέπουν με ικανοποίηση το έργο που θα αναπτύσσει σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης υπηρεσία αυτή με το προσωπικό της και πιστεύω ότι θα είναι πολύ θετική και η ε, ενδιάμεση επισκόπηση το 2013. Ιδιαίτερη σημασία δώσαμε στην επιμόρφωση, στην περαιτέρω κατάρτιση του προσωπικού, για την οποία προβλέψαμε ειδική διάταξη και επίσης ε, πάλι προερχόμενοι από διαφορετικές παραδόσεις υπόβαθρο θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν έτσι ώστε να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αυτή τη κοινή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Λίχτενμπέργκερ και τον κύριο Σάριου Φόλσκι για την κατάρτιση, τη βοήθεια που μα προσέφεραν στο θέμα τη κατάρτιση και τη ε, επιμόρφωση. Θα συνεχίσουμε φυσικά, θα τα ξαναπούμε τους επόμενους ε, μήνες και εβδομάδες και σας ε, διαβεβαίω ότι έχουμε πολύ μεγάλη σημασία αποδόσεις στην κατάρτιση αυτή. Επίσης, ως προς το κλίμα, το οικονομικό πάνω απ' όλα, στο οποίο ε, αναπτύσσονται αυτές οι προσπάθειες ε, τη ημέρων ημέρα. Είμαι υποχρεωμένη να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε ιδιαίτερα φιδωλοί στην αξιοποίηση των κονδυλίων και αποτελεσματικοί. Κυρίε και κύριοι, κάθε ε, Ευρωπαίος βλέπει καθημερινά τη σημασία του εθνούς εμπορίου, των διεθνών σχέσεων, της αντιμετώπισης τρομοκρατίας, έτσι λοιπόν θεωρώ καθήκον μου να εξασφαλίσω την αποτελεσματική και ικανοποιητική για όλους σας δράση αυτής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας, για την ε, παρουσίαση και παρακαλώ τώρα εκ μέρους του Συμβουλίου να λάβει το λόγο ο κύριος Ολυβίες Σαστέλ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωπε, κύριε Επίτροπε, κύριοι βουλευτές. Εξ ονόματος του Συμβουλίου επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους εισηγητές του Κοινοβουλίου οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά για τα διάφορα θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για την λειτουργία της ΕΓΕ, Γκρέσλε Ριβελίνη, για το δημοσιονομικό κανονισμό, ΡΑΠΚΑ για το προσωπικό και Γκουαλτιέρη και Σουριάν για τον διορθωτικό προϋπολογισμό. Μετά την πολιτική συμφωνία της Μαδρίτης και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 26 Ιουλίου ενέκρινε τη θέσπιση της ΕΙΕΔ. Για να μπορέσει όμως αυτή η υπηρεσία να λειτουργήσει έπρεπε να εγκρίνουμε αυτά τα τρία μέσα που προανέφερα. Οι εργασίες για τα διάφορα ντοσιέ ήταν πολύ σκληρές και στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν και σε επίπεδο κυρία Άστον και όλοι πραγματικά κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε ε, πρόθεσμα σε συμφωνία. Σήμερα λοιπόν εκφράζουμε τη χαρά μας, την ικανοποίησή μας για την ευόδοση αυτού του έργου. και μετά από την ψηφοφορία σε αυτήν εδώ την Ολομέλεια στις 25 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα εγκρίνει όλα αυτά τα μέτρα ούτως ώστε 1η Δεκεμβρίου να αρχίσει να είναι λειτουργική η υπηρεσία. Όλα τα έχουν πει η Λέντι Άστον, ε, οι εισηγητές, ο Επίτροπος. Εγώ το μόνο που θα κάνω είναι να τονίσω τον ιστορικό χαρακτήρα του γεγονότος. Ένα χρόνο μετά από την ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας πρόκειται για την πιο σημαντική της καινοτομία. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δηλαδή ενισχύονται οι διπλωματικές κοινέ δράσεις της Ένωσης. Βεβαίως τώρα αρχίζει το έργο και η πρόκληση πρέπει να είναι στο ύψος ε, των φιλοδοξιών μας. Εμείς βασιζόμαστε στη Λέδη Άρστον να αντιμετωπίσει αυτή την ε, πρόκληση και της εύχομαι καλή επιτυχία. Και για να ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε θέλω να ευχαριστήσω και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επικοδομητική του στάση και τη στράτευσή του που ήταν αποφασιστικές για αυτό το ντοσιέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Σαρουσβόλσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι από την Επιτροπή ΑΦΕΤ με μεγάλη πλειοψηφία είναι υπέρ ε, μιας δυνατής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης που να υφίσταται δημοκρατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο ε, που θα εκπροσωπεί την κοινότητα των 27 κρατών μελών, ε, που θα σέβεται την γεωγραφική κατανομή, την γεωγραφική διαφοροποίηση. Η ισορροπία γεωγραφική δεν ήταν στο παρελθόν σημαντική, ενώ είναι σήμερα και το, το 7 του ψηφίσματος και το άρθρο 6.6 το υπενθυμίζουν. Ε, έχουμε 200 από τις νέες χώρες εδώ και θα το παρακολουθούν αυτό. Υπάρχει γεωγραφική ισορροπία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην αρχική πρόταση, αλλά δεν είναι επαρκής. Βεβαίως ε, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την γεωγραφία επίσης, την ισότητα μεταξύ των φύλων. Οι άνδρες και οι γυναίκες είναι ίσοι. Μερικοί βεβαίω είναι πιο ίσοι από άλλους. Ελπίζουμε ότι οι διακρίσει θα διορθωθούν από εσά, Lady Ashton, σε αυτό που θα γίνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Φάρμ για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, ε, κυρία Άρστον, εκπρόσωποι του Συμβουλίου, υπήρξε η απόφαση της Μαδρίτης για τον προϋπολογισμό, αλλά για ορισμένα σημεία χρειάστηκε εμβάθυνση για μεγαλύτερη διαφάνεια, για μεγαλύτερη ευθύνη και πιο συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Πρόκειται για ένα εγγυημένο δικαίωμα στην πληροφόρησή μας για το συνολικό κόστος για τους ελέγχους πάνω στη διαχείριση ούτως ώστε να μην να, μην γίνεται, κρυφά η δράση αυτής της υπηρεσίας και όχι μόνο το κοινοβούλιο να είναι πληροφορημένο αλλά και ο απλός πολίτης να ξέρει τι κάνει αυτή η νέα υπηρεσία της Ένωσης. Πιστεύω ότι βάλαμε σήμερα τα θεμέλια που θα βοηθήσουν την Ένωση να ριζώσει στον κόσμο και να τον βελτιώσει με συμμετοχή των πολιτών. Ο κύριος Κάτσμαρεκ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Η χρωμαδότηση τη Επιτροπή Ανάπτυξη είναι θετική και ομόφωνα υποστηρίζουμε τις τροπολογίες που κατέθηκαν, ιδιαίτερα εκείνες που βαίνουν προς την κατεύθυνση της ε, επί τη βάση αντικειμενικών διαφανών ισότιμων διαδικασιών προσλήψεως του προσωπικού αυτή τη υπηρεσία. Αντίστοιχα δηλαδή με τι διατάξει που ισχύουν για το λοιπό προσωπικό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλες του κυρίου Ραπκάη, του κυρίου Συγητή για την ε, ε, στελέχωση τη υπηρεσία που προκύπτουν κατόπιν πολιτική συμφωνία, ιδιαίτερα προ την ισότιμη μεταχείριση των δύο φύλων και καταγωγή και ισότιμης κατανομής μεταξύ προσωπικού προερχομένου από τις ευρωπαϊκές ε, υπηρεσίες και τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών μας ε, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει πολύ ικανοποιητικά αυτή η υπηρεσία και ελπίζουμε ότι θα αναγνωρίσει τη σημασία της αναπτυξιακής συνεργασίας η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ώστε αυτή να μην μετατρεπεί μόνο σε ένα είδους δέλεαρ ε, μόνο αλλά να είναι ουσιαστική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Άστον. Πολλοί από την ομάδα μου θέλουν Πολλοί από την ομάδα μου θέλουν να υπάρχει μια γεωγραφική ισορροπία και ισορροπία φίλων στην ΕΕΔ. Αλλά θέλουμε να σταματήσουμε τη ρουσφετολογία και τις διάφορες εθνικές οικολογικές ε, σταυροφορίες. Θέλουμε να υπάρχει αξιοκρατία. Καταλαβαίνουμε όμως ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε κατευθείαν στο καλό αποτέλεσμα. Θα τα καταφέρουμε με το χρόνο. Ξέρουμε όμως ότι αν δεν, κυρία αν δεν πετύχουμε την ισορροπία που θέλουμε, αυτοί που θέλουν να σας κάψουν το λάκκο, κυρία Άστον, θα, τη δράξουν αυτή την ευκαιρία και θα τα καταφέρουν. Η ομάδα μου σας υποστηρίζει και τρέφει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας. Πρέπει να, δώσουμε, ε, να σας δώσουμε τα μέσα να τα καταφέρουμε και να πετύχουμε την ΕΙΕΔ. Αν εσείς όμως σε δύο χρόνια έρθετε και μας πείτε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην κατανομή των συνεργατών σας, σίγουρα θα προκύψει ένα πρόβλημα στην απαλλαγή. Καλώς, καλή σας τύχη. Ο κύριος Σαρίφ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, επιτέλους ε, καταλήγουμε ε, στο τέλος όλης αυτής της διεργασίας για τις βάσεις της ΕΙΕΔ. Θέλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε τους εισηγητές ε, για την ποιότητα της εργασίας τους. Θέλουμε να αναπτυχθεί μια πραγματική ευρωπαϊκή διπλωματία η οποία δεν θα αποτελεί απλώς το σύνολο των διπλωματικών υπηρεσιών των κρατών μελών. Γι' αυτό ο προϋπολογισμός που δίνουμε σήμερα πρέπει και τα κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά ούτως ώστε να έχουμε μια συνοχή των εξωτερικών πολιτικών της Ένοχης. Η εμπορική πολιτική δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητες ε, της, ΥΠΑ, της ε, κυρίας Άστον, αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξει σωστός διάλογο με τον, με τον ομόλογο της ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσα από την εξωτερική πολιτική να έχουμε προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εμπορικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες. Θέλουμε λοιπόν να βαρύνουμε στην ε, στο διεθνές πολιτικό προσκήνιο με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα προσωπικά να υποστηρίξω το Γκρέσλε Ριβελίνη και τον κύριο Ραπκά για την εξαίρετη εργασία είναι σαφές για μας ότι βεβαίως πρόκειται για μια διαδικασία περίπλοκη η υπηρεσία εξωτερικής δράσης όπου θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα και την εκπροσώπηση των κρατών μελών. Ταυτόχρονα η υπηρεσία πρέπει να είναι δυνατή και η Ευρώπη στην διεθνή ε, σκηνή να γίνει μεγάλος ο πρωταγωνιστής η πρόταση για γεωγραφική ισορροπία που ε, ψηφίστηκε με πλειοψηφία στην ΑΦΕΤ και στην Επίτροπη Ανάπτυξης και που συμφωνεί με το ψήφισμα της 8ης Ιουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αντανακλάται στην έκθεση ΡΑΠΚΑ. Γι' αυτό στρέφομαι σε εσά, λέει Διάστον, διότι εσείς είστε το άτομο που έχει συμφέρον ε, για την κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να είναι πίσω σας, να είναι στο πλευρό σας. Γι' αυτό θα ήθελα ε, να διασφαλίσετε την ε, γεωγραφική ε, ισορροπία. Καλή τύχη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού θέλω να χαιρετήσω αυτή την εισήγηση και αυτή την υπηρεσία εξωτερικής δράσης που είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την υπηρεσία αλλά είναι σημαντικό να θέσουμε τις βασικές αρχές οι οποίες στο μέλλον θα ισχύσουν για αυτήν την γραμμή του προϋπολογισμού. Είχαμε πολλές συζητήσεις ε, με τον Γενικό Διευθυντή της Εξωτερικές Υποθέσεις, αλλά το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θα πρέπει οι κανόνες να είναι σαφείς, να μην υπάρχουν επικαλύψεις και να είναι όλα σαφή και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των κονδυλίων. πρέπει η εργασία, η απόδοση να είναι αποτελεσματική. Αυτή είναι η μεγάλη προτεραιότητα. Τα κονδύλια θα έρθουν από τρει πηγέ. και ε, το προσωπικό θα προέρχεται από την Επιτροπή, από το Συμβούλιο και από τα κράτη-μέλη, από τρει πηγέ. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία στο σώμα αυτό των ανδρών και των γυναικών. Χρειαζόμαστε εκπαίδευση για το μέλλον και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης θα πρέπει να ελέγχονται ε, κάθε χρόνο. κύριος Μπελτσίτους ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, επίτροποι, εκπρόσωποι του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους εισηγητές που κατόρθωσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιτύχουν πολιτική συμφωνία με τα άλλα θεσμικά όργανα και να θέσουν τα θεμέλια για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Η υπηρεσία αυτή θα συμβάλλει στο υψηλότερο επίπεδο στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής της ασφάλειας και θα ενισχύσουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή εικονίστρα. Θα πρέπει να ε, τηρήσουν ε, τις αρχές της ε, καλής διαχείρισης. Έχουμε 9,5 εκατομμύρια ευρώ για την υπηρεσία, αλλά θα, μετά το πρώτο έτος θα υπάρξει αξιολόγηση όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει τον οικονομικό απολογισμό. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπεύθυνο ρόλο για την λειτουργία ε, της υπηρεσίας για την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων και για να υπάρχει μια καλή προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο και τους λαούς. Γεύκα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρία Άστον. Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, ε, όλοι μας δεν αμφιβάλλουμε για τη σημασία της ε, λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, και η εργασία μας τους τελευταίους μήνες έχει βασιστεί στην, στο θέμα αυτό. Εργαζόμαστε σε δύσκολους καιρούς, αλλά τελικά καταλήξαμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και ελπίζω ότι ο συμβασμός που επιτεύχθηκε θα μπορέσει να οδηγήσει σε θετικά αποτέλεσματα στο τέλος η Επιτροπή ε, κατέθεσε τροποποιήσεις για τον κανονισμό ε, του προσωπικού, τόσο ώστε η υπηρεσία να είναι ανεξάρτητη και να έχει τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες που χρειάζεται. Νομίζω ότι οι τροπολογίες που κατατέθηκαν εχθές το εγγυώνται αυτό. Βέβαια δεν είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι με αυτές τις τροπολογίες, κυρίως για ένα θέμα, το θέμα της γεωγραφικής ισορροπίας που θα μπορούσε να προβλέπετε καλύτερα στο κείμενο, να εξασφαλίζετε καλύτερα. Ελπίζω, είπατε εκπρόσωπος, να λάβει υπόψη ε, το θέμα αυτό, ούτως ώστε όλα τα κράτη-μέλη να εκπροσωπούνται καλά στην υπηρεσία και ελπίζω ότι θα μας αναφέρετε ε, τις διάφορες δράσεις ε, της υπηρεσίας. Η διπλωματία μας πρέπει να είναι ευρωπαϊκή και θα πρέπει ε, βεβαίως δεν θα έπρεπε να είναι σημαντική η εθνικότητα των εργαζομένων στην υπηρεσία αλλά οι ρίζες μας είναι σημαντικές και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Βεβαίως υπάρχουν κρατημέλη που υποεκπροσωπούνται σε όλα τα θεσμικά όργανα. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε ε, διαφορετική αλλά και ενωμένη ε, πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε γεωγραφική ισορροπία που να περιλαμβάνεται στο κείμενο, να αναφέρεται στο κείμενο. Δεν πρόκειται για ποσοστώσεις για τα κράτη-μέλη αλλά για γεωγραφική ισορροπία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συγγιστές για την αγαστή συνεργασία. Ελπίζω ότι η Λέιδη Άστον θα χρησιμοποιήσει καλά τη συνεργασία μας στο μέλλον. Ο κύριος Σβόποντα, δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ήθελα θερμά να ευχαριστώ τους συζητητές για το έργο τους και για τις συμβαστικές λύσεις που οποίες μπορούσαν να καταλήξουν. Φυσικά, ίσως να μην όλοι ικανοποιημένοι 100%. Αντιλαμβάνομαι και τα μελήματα για την εκπροσώπηση των φίλων, τη γεωγραφική εκπροσώπηση, που θα πρέπει να απασχολεί όχι μόνο ε, τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου αλλά όλα τα μέλη, όλους τους βουλευτές όπως επίσης πρέπει να περιμένουμε με όλη για ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο προσωπικό αυτής της υπηρεσίας. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Έχουμε να κάνουμε με την ανάγκη να δημιουργηθεί μια υπηρεσία ύψης της ποιότητας. Και είναι η ώρα πλέον να λάβουμε δράση, είναι η ώρα να δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να, εκπροσωπήσουμε, να εξασφαλίσουμε την εκπροσώπηση Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή σκηνή. Κυρία Άστον, έχει αναλάβει αυτό το καθήκον. Βλέπουμε και ελπίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Και Φερρυπίν στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να πείσουμε όχι μόνο τους ε, εμπλεκόμενους αλλά όλους τους παράγοντες ε, ώστε να αναγνωριστεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τις Ηνωμένε Πολιτείες όταν έχουμε να διαπραγματευτούμε ζητήματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Τα διαπραγματευόμαστε από κοινού. Είτε πρόκειται για τρομοκρατία, είτε πρόκειται για αντιμετώπιση των συνεπειών τη παγκοσμιοποίηση. Όταν έχουμε να κάνουμε με την Κίνα, νέε αναδυόμενε δυνάμει, νέα αναδυόμενη δύναμη μάλλον στον κόσμο, θα πρέπει να είμαστε θέση να αντιμετωπίσουμε και ζητήματα εθνικισμού και μιας κάποιας ε, επιθετικότητας που αναπτύσσει η Κίνα στην περιφέρεια της και να είμαστε θέση ως ισότιμοι εταίροι να συνομιλούμε τα ζητήματα αυτά. Και θα πρέπει να είμαστε σε θέση μέσα σε, στους μεγάλους πολυμερείς οργανισμούς να έχουμε εκπροσώπηση και ισχυρή παρουσία ώστε να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεκτή ως παγκόσμιος παράγων στη διεθνή σκηνή. Αυτά είναι όλα καθήκοντα που θα πρέπει να επομιστεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσεω. Επίση, η Προεδρία, και εσεί το αναφέρατε κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, υποστηρίζει την ΕΕΔ. Ελπίζω ταυτόχρονα ότι θα της επιτρέψετε να ανοίξει τα φτερά της και να αναλάβει δράση χωρίς να παρεμποδίσετε τις επιλογές της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Η κυρία Βίξτρομ έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Πρώτα απ' όλα κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτήν την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ όλων όσων συνεργάστηκαν για το θέμα. Η κυρία Άστον δεν είχε καθόλου εύκολες, ε, ε, εύκολη δουλειά στο να μπορέσει να προχωρήσει δηλαδή στη σύσταση της ΕΕΔ. Πάντως ε, σήμερα έχουν στηθεί βάσεις για να έχουμε μια πραγματικά αποτελεσματική και αντιπροσωπευτική οργάνωση που θα εκπροσωπεί την Ευρώπη, τις αξίες της και τα συμφέροντά της ανά τον κόσμο, ενισχύοντας ε, την ευρωπαϊκή διαφορετικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από άτομα με διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα και εμπειρίες. Οι υπάλληλοι των εξωτερικών υπηρεσιών θα προσληφθούν από όλα τα κράτη-μέλη και αυτό αποτελεί και το σημείο δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε σε αυτήν τη νέα υπηρεσία να είναι οι αξίες και οι γνώσεις που θα πρέπει να υπερισχύσουν. Το ρητό του Κοινοβουλίου είναι ενωμένη στη διαφορετικότητα. Πρόκειται για ένα ρητό με ένα πολύ βαθύ νόημα. Ελπίζω η εξωτερική υπηρεσία από την αρχή κυρία Άστον να λειτουργήσει ως πραγματική υπηρεσία που θα εκπροσωπεί τη διαφορετικότητα όλων των κρατών μελών και όλους τους πολίτες των κρατών μελών άντρες και γυναίκες. Πρέπει να προωθήσουμε την κατάρτιση σε όλα τα κράτη-μέλη αγοριών και κοριτσιών ούτως ώστε να θέσουν υποψηφιότητα για να γίνουν υπάλληλοι σε αυτήν την υπηρεσία. Μπράτνερ, μισή λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για τα όσα πράξαμε, για τα όσα επιτύχαμε μέχρι σήμερα. Προσδορίσαμε τι προτεραιότητε, διαφυλάξαμε τι επιλογέ Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δυνατότητα ε, δημοσιονομικού ελέγχου, ιδιαίτερα με το διορθωτικό προπολογισμό. Έχουμε επίση εξασφαλίσει μια βάση ισότιμη λειτουργία μέσα σε πνεύμα αγαστή συνεργασία για αυτήν την υπηρεσία εξωτερική ε, δράση με μέτρα ενσωμάτωσης, ε, ισότιμης μάλλον μεταχείρισης των δύο φύλων και, της, και ισότιμη γεωγραφική εκπροσώπηση. Ναι, όλα αυτά τα καταφέραμε. Έχουμε όμως επιτύχει την δημιουργία μιας σύγχρονης διπλωματικής υπηρεσίας που να μην αποτελεί απλώς το συνονθήλευμα ή το άθροισμα καλύτερα 28 διαφορετικών διπλωματικών υπηρεσιών. Τι έχουμε ακόμα να κάνουμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Χρειάζεται ένας αποτελεσματικός συντονισμός στους διάφορους τομεί ε, της πολιτικής. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Δεύτερον, Πρέπει να ενισχύσουμε την διαχείριση των κρίσεων και την πρόληψη των συγκρούσεων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα με την κατάλληλη δράση όπως ονομάζεται και τη δημιουργία νέων θέσεων που μπορούν να αναπτυχθούν σε συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής. Μέσα λοιπόν στην ευθεία αυτή χρειαζόμαστε περισσότερους ε, πρέσβεις Β. Χρειαζόμαστε, κυρία Άστον, διπλωμάτης του 19ου αιώνα σε αυτή τη σύγχρονη υπηρεσία. Δεν χρειάζεται να μπορούμε κυρία Άστο να βρούμε τους ανθρώπους που πραγματικά χρειαζόμαστε για τη δουλειά που τους χρειαζόμαστε. Ελπίζω λοιπόν το οργανόγραμμά σας και οι προτεραιότητές σας να προσδιορίζουν ακριβώς αυτούς τους στόχους και να εξυπηρετούν αυτούς τους στόχους έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε περισσότερα από ότι μια εθνική διπλωματική υπηρεσία και διαχείριση κρίσεων και πρόληψη συγκρούσεων. Μια ιδιαίτερη μονάδα Φερρυπίν ή στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα των ανθρωπινών δικαιωμάτων και σύγκριση στο επίπεδο το σχετικό δυναμικό. Και επίση η ισότητα των φύλων δεν εξασφαλίζεται μόνο με το πόσο ανθρώπου θα προσλάβουμε από το κάθε φίλο, αλλά με την ενσωμάτωση τη θέση των φύλων σε κάθε ζήτημα πολιτική που θα χαράσει η υπηρεσία σα. Και παρακαλώ αυτό να λαμβάνετε υπόψη και στην ε, ανασκόπηση παρελθουσών δράσεων ε, εξωτερικών σχέσεων της ΚΕΠΑ δηλαδή αλλά και στο παρόν και το μέλλον. Και ελπίζω να έχετε πολύ καλή και επικοδομητική εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος για ένα λεπτό. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση 27 κρατών μελών. Αυτό πρέπει να αντανακλάται επίση στην διαμόρφωση ενός οργάνου που θα μας εκπροσωπεί προς τα έξω. Μερικοί μπορεί να πιστεύουν ε, ότι δεν τη χάνουν της καλής μεταχείρισης από τη νέα υπηρεσία ορισμένες χώρες, η οποία θα έπρεπε να αντανακλά τις διαφορετικούς πολιτισμούς ε, και παραδόσεις των διαφόρων χωρών. Γι' αυτό καταθέσαμε ψηφίσαμε μια τροπολογία που να εξασφαλίσει στο κείμενο γεωγραφική ισορροπία ε, ούτω ώστε σε περίπτωση ισοτήμων αρμοδιοτήτων και προσόντων των υποψηφίων να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο το γεωγραφικό. Βεβαίως δεν πρέπει το κριτήριο αυτό να είναι άκαπτο αλλά να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο συμπληρωματικό κριτήριο ούτω ώστε να διορθωθεί η έλλειψη ισορροπίας που υπάρχει στο κείμενο και ούτω ώστε στο μέλλον να υπάρχει καλύτερη γεωγραφική κατανομή. Βεβαίως τα προσόντα είναι το σημαντικότερο ε, διότι ώστε να λειτουργήσει καλά η υπηρεσία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάιερ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχήν να κάνω να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου σήμερα λέγοντας ότι η Γκούε εκφράζει την αλληλεγγύη της με τους εργαζόμενους της Γαλλίας οι οποίοι διαμαρτύρονται για την αντιδραστική πολιτική του κυρίου Σαρκοζή. Ο πρόεδρος είπε προηγουμένως ότι θα, να θα αργήσουν να έρθουν οι αρμόδιοι λόγω καθυστερήσεων. Λοιπόν, οι καθυστερήσεις έχουν ένα όνομα και είναι οι απεργίες. Εγώ λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη δουλειά τους, αλλά πρέπει να τους πω ότι σήμερα η ομάδα μου θα κάνει αποχή διότι δεν πετύχαμε αυτό το οποίο εμείς θέλαμε, δηλαδή τον εξαντλητικό έλεγχο εκ μέρους του Κοινοβουλίου της ΑΕΕΦ και η διάρθρωσή της εμάς δεν μας πείθει. Δηλαδή που θα αναλαμβάνει τις πλήρεις, θα καλύπτει τις πλήρεις πτυχές της ΚΕΠΑ. Εμείς δώσαμε μία μεγάλη δημοκρατική μάχη εκ μέρους της ομάδας μας για τον απόλυτο έλεγχο της πτυχής ε, της ασφάλειας. Θέλαμε λοιπόν το θέμα της ασφάλειας να περάνει μέσα από τον απόλυτο και εξαντλητικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Κάτι τέτοιο δεν το πετύχαμε. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν θα ψηφίσουμε αύριο. Πάντως ευχαριστώ για τη δουλειά που έγινε μέχρι τώρα. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους στην ε, Γαλλία. Ο Προβέρα. Στον ορισμό της νέας διπλωματικής υπηρεσίας δεν πρέπει να, να, να, επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Πρέπει να έχουμε ένα ευέλικτο, ένα ευέλικτο οργανόγραμμα και αποτελεσματικό. Δεν θα πρέπει να επιλέγονται οι υπάλληλοι λόγω της γεωγραφικής τους προέλευσης ή λόγω του φίλου τους. Μόνο λόγω της ποιότητάς τους. Σίγουρα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν εκπροσώπηση στο υπαλληλικό οργανόγραμμα της ε, υπηρεσίας και θα πρέπει να υπάρχει και γυναικεία εκπροσώπηση. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της αξιοκρατίας και της αριστείας. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ίση, ίσα δικαιώματα πρόσβαση στη σταδιοδρομία για όλους, χωρίς διακρίσεις. Ε, για την κατάρτιση έχουμε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, το οποίο έχει και την εμπειρία της κατάρτισης. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι άχρηστο το και δαπανηρό το να οικοδομήσουμε εκ νέου μια νέα Ευρωπαϊκή Ακαδημία. Η ε, κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι συνάδελφοι. για να μπορέσουμε να εκπροσωπούμε, για να μπορέσει να εκπροσωπεί η ΕΕΔ αποτελεσματικά τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ τα έξω, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να εκφράζει με μία φωνή τι θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή τα πολιτικά όργανα, τα πολιτικά εργαλεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενοποιημένα μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο και επαναπροσδιορισμένα όπως αναφέρεται σε εκθέσεις των συναδέλφων, πρέπει εν ώψη αυτής της ε, καινοτόμων δομής που αναπτύσσεται να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις διαφάνειας της ε, λογοδοσίας και της διαφανούς διαχείρισης των δημοσιονομικών, έτσι ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά αυτή η δράση. Όμως χρειάζεται και το προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να ε, διατεθεί στην υπηρεσία αυτή η διάρθρωση της υπηρεσίας ως τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ενσωμάτωσή της μέσα στο δημοσιονομικό κανονισμό σημαίνει ταυτόχρονα την υποχρέωση της ε, διαφάνειας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη διαδικασία της απαλλαγής, την οποία όλοι θα μεριμνήσουμε να ε, φέρουμε σε σιωπέρας. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι το προσωπικό θα πρέπει να επιλέγεται με βάση αξιοκρατικά κριτήρια και δεν αρκεί να λέμε ότι χρειάζεται να έχουμε ισότιμη εκπροσώπηση και των γυναικών. Πρέπει να βρούμε καλά καταρτισμένε γυναίκε. Υπάρχουν τέτοιε γυναίκε, αρκεί να τι βρούμε. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριο Μπροκ. Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο Φρανκ Σινάτρα επωνομαζόταν The Voice, αλλά χωρίς μια big band πίσω του δεν ήταν τίποτα. Ε, εσείς κυρία Άστον τώρα είστε η φωνή της Ευρώπης και από πίσω σας με τη μορφή αυτής της εξωτερικής υπηρεσίας έχετε την ορχήστρα η οποία σε αρμονία θα μπορέσει να προβάλλει τα, την Ευρώπη, τις θέσεις της και πάνω απ' όλα να εξασφαλίσει σαν δεύτερο βήμα, για το πρώτο βήμα στην Ευρώπη ήταν η εξασφάλιση εσωτερικής ειρήνης στα όρια δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα σε δεύτερο βήμα να προχωρήσουμε στις, ε, στην ανάπτυξη των πνευματικών σχέσεων, στην καταπολέμηση τρομοκρατία, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της παγκοσμιοποίησης. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα το οποίο έχετε να πραγματοποιήσετε με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, με πολλή δουλειά και βέβαια ως επικεφαλής αυτής της ορχήστρας θα και εσείς κυρία Άστον. Ο έλεγχος η δημοσιονομική εποπτεία από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φυσικά ε, συμπληρώνουν αυτή την εικόνα και εξασφαλίζουν καλή λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης με ένα καλό προσωπικό το οποίο θα επιλεγεί και πιστεύω ότι μπορέσαμε εμείς να ενισχύσουμε τη διάσταση τη γεωγραφική και τη ισότιμη αντιμετώπιση των φύλων ή ενσωμάτωση των φύλων, αντίθετα από ό,τι έκανε το Συμβούλιο. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι Εάν καταφέρει αυτή η υπηρεσία πράγματι να έχει τη γεωγραφική εκπροσώπηση, την εκπροσώπηση των φίλων όπω την επιθυμούμε, αυτό το οφείλει σε εμά, τι προσπάθειε του Κοινοβουλίου. Και κυρίε και κύριοι, έχουμε να κάνουμε με ένα μέσον το οποίο πρέπει να αφήσουμε να λειτουργήσει αποτελεσματικά μεν, με ευελιξία μεν, αλλά ταυτόχρονα και με αυστηρό έλεγχο δε. Και κύριε Άστον, σα διαβεβαιώ ότι θα ακούσετε και πολλέ επικρίσει από πλευρά μα όταν και εάν δεν συμφωνούμε με τι επιλογέ σα στο θέμα αυτό μπορούμε όλοι και μόνο όλοι από κοινού να προσδιορίσουμε αυτό που πράγματι θέλει ο πολιτή ω εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σεβερίν, παρακαλώ. There will be no any δεν θα υπάρχει καμία επιτυχία στην Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη χωρίς οξυδέρκεια για το πόσα θα πρέπει τα κοινά μας συμφέροντα να προωθηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε φιλόδοξη ε, υπηρεσία αποτελεσματική που δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς ένα προσωπικό ε, που να βασίζεται στην αξιοκρατία η πρόσληψή του. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε για αυτές τις αρχές, αλλά ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες και είναι ακριβώς αυτές οι λεπτομέρειες που μεταμορφώνουν μια έκθεση που θα ήταν τεχνική σε μια πηγή εμπαθούς συζήτησης που επιφέρει διχόνοια. Βεβαίως, έχουμε, ε, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει θέμα ποσοστώσεων μεταξύ παλαιών και νέων χωρών. Ε, η ε, τον, για να έχουμε μια καλή κοινότητα και ένα κοινοτικό ε, πνεύμα πρέπει κάθε χώρα να ε, σκέφτεται ότι έχει την σωστή μεταχείριση βάσει της αξιοκρατίας, βάσει των αξιών της, των ε, χαρακτηριστικών τους. Νομίζω ότι ο Θεός έχει κατανείμει με αξιοκρατικό τρόπο τα διάφορα χαρακτηριστικά ανάμεσα στους δυτικούς, στους ανατολικούς, στους άνδρες, στις γυναίκες, στις μεγάλες και στις μικρές χώρες. Μερικοί στην η Ευρωπαϊκή μας Ένωση, κυρίως από τις νέες χώρες, αλλά όχι μόνο, αισθάνονται ότι είναι αντικείμενα διακρίσεων, θύματα διακρίσεων. Πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη με πάρα πολύ προσοχή τα κριτήρια δεν αμφισβητούνται αλλά αμφισβητείται η έλλειψη εξασφάλισης ότι ε, θα υλοποιηθούν σωστά και ότι θα υπάρξουν ανισορροπίες. Ελπίζω είπατε, η εκπρόσωπος να διορθώσει στην πορεία αυτές τις στρεβλώσεις, αυτές τις ανισορροπίες και ελπίζω ότι η μελλοντική διπλωματική ακαδημία ή δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε ένα σώμα Ευρωπαίων διπλωματών που θα είναι ε, πιστοί ε, στις κοινέ μας αρχές, στα κοινά μας συμφέροντα και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν τέλειο. Τέλειο, Άντριαν. Ο κύριος Γκμπράντι, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση αναφέρεται κυρίως στην εποπτεία στον έλεγχο της υπηρεσίας αυτής, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την σημασία της υπηρεσίας αυτής. Είναι πολύ μεγάλη η σημασία της υπηρεσίας, είναι ένα από τα πρώτα βήματα προς μια πολιτική ευρωπαϊκή εξωτερική. Η χώρα μου έχει, ε, ήταν πολύ συχνά εσωστρεφής. Βλέπουμε ότι ε, αναφέρεται η υπηρεσία αυτή στην ε, συμφωνία την διακυβερνητική. Πρόκειται για κάτι το περιορισμένο για την ώρα, αλλά σύντομα η υπηρεσία αυτή θα μπορέσει να ασχοληθεί με έργο πολιτικό εξωτερικής πολιτικής. Μιλάμε σήμερα για τη χρηματοδότηση και οργάνωση της υπηρεσίας αυτής. Είναι σημαντικό αυτό. Η ευθύνη, η αρμοδιότητα, η χρηματοοικονομική και η διαφάνεια είναι ουσιαστικά θέματα για την επιτυχία της υπηρεσίας αυτής. Χαίρομαι για τη συμφωνία που βρέθηκε μεταξύ των θεσμικών οργάνων, διότι υπήρχε μια απειλή και ως Κοινοβούλιο παρουσιάσαμε διεκδικήσεις, απαιτήσει ε, λεπτομερείς. Θα ήθελα να συγχαρώ λοιπόν τους εισηγητές. Το πακέτο αυτό είναι ένα καλό πακέτο και οι συναδελφοί μου θα το εγκρίνουν και ελπίζω ότι μετά την αυριανή ψηφοφορία η υπηρεσία αυτή θα μπορέσει χωρίς καμία καθυστέρηση να αρχίσει τις εργασίες. Ο κύριος Τάνο, ένα λεπτό. Πρόεδρε, μια υβριδική σου η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση έχει απασχολήσει το Κοινοβούλιο με πολλέ συζητήσει και μη τι άλλο η κυρία Άστον άξιε συγχαρητηρίων γιατί μέσα σε μία περίοδο κρίση στην ε, ζώνη του ευρώ ασχολούμαστε με την υπηρεσία τη. Ίσως με τον τρόπο αυτό μπορέσουν να περικόψουν ε, κάποιοι τη δυνατότητα της ε, Μεγάλης Βρετανίας να αναπτύσσει αυτόνομη εξωτερική δράση, αυτόνομη δηλαδή διπλωματία, αλλά εμεί θα μεριμνήσουμε είτε Πρόκειται για το λόμπι των Βρετανών ε, υπηρεσιών, των Βρετανικών υπηρεσιών και των Βρετανών ε, διπλωματών σε εκπροσώπηση των, υπηρεσία της υπηρεσίας γιατί είναι υποεκπροσωπούμενη η Μεγάλη Βρετανία στις γλυπές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε διαφυλάσσοντας την αρχή της αξιοκρατίας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν και υπερβολικές δαπάνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να την ευήκονουν στην ανάγκη για ε, λιτότητα και ιδιαίτερα στον προπολογισμό αυτής της υπηρεσία όπου η εξωτερική της δράση πρέπει να εξασφαλίσει εμπιστοσύνη, αξιοπιστία ενώπιον του Ευρωπαίου πολίτη με την φιδωλή διαχείριση. Κύριε Τάνοκ, είπατε εσεί ότι το, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται, αλλά φαντάζομαι θα το Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι. Πρόεδρο. Απλώ για να διευρύνουμε κάπω την πρόπτικη, το ανέφερα. Ο κύριο Μαστάλκα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ΕΕΔ αποτελεί ένα νέο μέσο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας για την θεσμοθέτηση των εξωτερικών δράσεων της Ένωσης. Αλλά η δημιουργία αυτής της υπηρεσίας συνοδεύεται από διάφορες προβληματικές. Η πολιτική άμυνας είναι πάντοτε αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επίσης υπάρχει πάντοτε το δικαίωμα βέτο ας πούμε δείτε για τη συμμετοχή στον πόλεμο του Ιράκ ε, ή στο Κωσυφοπαίδιο όπου δεν υπήρξε μια κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εξωτερικά θέματα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πλήρη ατζέντα και να λαμβάνει κανείς υπόψη ότι οι αποφάσεις οι οποίες θα λαμβάνονται πρέπει να είναι αποφάσεις όλων των κρατών μελών και να υπάρχει εκπροσώπηση των νέων κρατών μελών. Η κυρία Αντρέασεν. Η ιδέα για μια εξωτερική, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση δεν ήταν ε, ποτέ ευπρόσδεκτη στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω η γραφειοκρατία μπόρεσε να πουλήσει αυτό το, αυτή την ιδέα, υποσχόμενη ότι θα είναι ουδέτερη δημοσιονομικά. Βλέπουμε όμω ότι δεν θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, ούτε καν θα περιοριστεί στα 441 εκατομμύρια ευρώ που είχαν αρχικά προβλεφθεί, θα κοστίσει επιπλέον 34 εκατομμύρια ευρώ. Η σημασία λοιπόν του δημοσιονομικού κανονισμού που ζητεί ε, λογοδεσία από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του εσωτερικού δημοσιονομικού ελεγκτή ε, σημαίνει αντίθετα από ό,τι συμφωνηθεί στην Μαδρίτη, ότι δεν είναι ανεξάρτητη αυτή η υπηρεσία δημοσιονομικά με δικό της ανεξάρτητο δημοσιονομικό ελεγκτή, εσωτερικό ελεγκτή, πράγμα το οποίο δεν είχε συμφωνηθεί στη Μαδρίτη και τελικά παρετούμεθα από αυτές τις συμφωνίες και προχωρούμε σε μια θάλασσα αβεβαιότητας και σύγχυσης. Είναι τροπή αυτή η προεξέλιξη. Πρέπει να πω ότι δεν εκπλήσουμε. Βλέπω όμως ότι όπως πάντα ο Ευρωπαίος Φορολογούμενος θα πληρώσει τα σπασμένα αυτής αναποτελεσματικότητας. Ευχαριστώ κύριος Χάρτονγκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, μιλάμε για χρηματοδότηση μιας νέας υπηρεσίας. Είναι λυπηρή ημέρα αυτή, ενώ οι Ολλανδοί αποφάνθηκαν για την συνθήκη της Λισαβόνας και σήμερα με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε αυτή την υπηρεσία που θα είναι μια γραφειοκρατία που θα κοστίσει πάρα πολύ ακριβά. Το πολιτικό λόμπι κοστίζει ακριβά των ευρωκρατών αλλά δεν αποφέρει τίποτα. Ε, δεν θα συμφωνήσουμε για να δώσουμε χρήματα σε αυτήν την υπηρεσία. Λέμε όχι σε αυτή την υπηρεσία, λέμε όχι στο ευρωπαϊκό υπερκράτος. Ναι ε, για την δημοκρατία και την αλήθεια των κυρίαρχων κρατών. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συζητούμε εδώ για την ομορφή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσεων. Δεν μπορούμε να ξεχνούμε την γεωγραφική ισορροπία στην σύνθεση του προσωπικού της υπηρεσίας αυτής. Για την ώρα ο αριθμός των ατόμων από τα 15 κράτη-μέλη, τα παλιά κράτη-μέλη είναι πολύ ψηλότερος ο αριθμός, σημαντικά υψηλότερος από ό,τι τα άτομα από τα νέα κράτη-μέλη. Μερικά στατιστικά στοιχεία είχαμε δύο πρέσβεις από νέες χώρες, από πάνω, μεταξύ πάνω από 100 πρέσβευτών. Και η ομάδα των, στην ομάδα των 29 νέων πρεσβευτών έχουμε μόνο δύο από νέες χώρες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ένας κανόνας ε, για τη νέα υπηρεσία εξωτερικής δράσης αν δεν εξασφαλίσουμε καλή ισορροπία και γεωγραφική εκπροσώπηση. Δεν μπορούμε να έχουμε μια σύγχρονη υπηρεσία εξωτερικής δράσης που θα λειτουργεί για την προστασία των συμφερόντων όλων μας και δεν θα μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι ε, για την ποιότητα μιας τέτοιας υπηρεσίας Ελπίζω η μεταβετική ε, περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας έχουμε υποεκπροσώπηση κρατών μελών ε, θα ε, λήξει αυτό που θα μπορούσε να είναι μια λύση ούτως ώστε να φτάσουμε σε κάποια χρονική στιγμή όπου θα εξασφαλιστεί η γεωγραφική ισορροπία και ισότητα και τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μια πραγματική φωνή στη διεθνή κονίστρα. Ευχαριστώ. Κύριος Βίτζενεν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συναδελφοί. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που εδώ στο Κοινοβούλιο συζητούμε τη δομή και τη χρηματοδότηση, το γενικό πλαίσιο δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Από αύριο που θα ψηφίσουμε, μπορούμε να περιμένουμε συγκεκριμένα πια αποτελέσματα. Όπως δείχνει σήμερα η συζήτηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταστεί το θεσμικό κοινό όργανο το οποίο θα μπορεί να δίνει όθηση, ιδέες, στήριξη στην ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Έτσι ώστε να καταστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ορατή στη διεθνή σκηνή. Είναι ίσως το πιο απτό αποτέλεσμα της συνθήκης Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Όλοι πιστεύω θέλουμε να δούμε την επιτυχή της ολοκλήρωση στην κυρία Άστον, θα ήθελα να πω ότι όταν ανέλαβε, όταν διορίστηκε μάλλον ε, ως είπατε εκπρόσωπος, άκουσε πολλές επικρίσεις και από εφέτος που ανέλαβε καθήκοντας είπατε εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η μόνη εκπρόσωπος εξωτερικής υπηρεσίας που εκπροσωπούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γεωγραφική ε, καταγωγή και η ισότιμη εκπροσώπηση, λένε πολλοί συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντική. Ναι, αλλά με αξιοκρατία. Και γι' αυτό πιστεύουμε, κύριε Άστον, ότι η δική σας στράτευση και αποφασιστικότητα θα είναι κρίσιμη σημασία για την επιτυχή ε, λειτουργία της υπηρεσία. Ο κύριος Λάμπστορφ. Πρόεδρε, έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα απτό αποτέλεσμα της συνθήκης Λισαβόνας και η κυρία Άστον πλέον δεν είναι η ε, Υπουργό Εξωτερικών εν το γίγνεσθε του υποκατασκευήν Υπουργείου Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η πραγματική Υπουργό Εξωτερικών του πραγματικού Ευρωπαϊκού Υπουργείου των Εξωτερικών. Κλείνει έτσι μια περίοδο αντιπαραθέσεων. Ε, πέρυσι το χρονοτούπολο από τι ιστορία στην παλαιά ΚΕΠΑ προχωρούμε προ ουσιαστική λειτουργία μια εξωτερική υπηρεσία με δημοσιονομικό έλεγχο, με πνεύμα συνεργασία με δημοκρατικό έλεγχο. Γεωγραφικές ποσοστώσεις δεν θα υπάρξουν. Φαίνεται ότι ενδιαφέρει πολλού το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει ε, γεωγραφική ποσόστοση και πρέπει να πω ότι ενώ η Γερμανία θα ήταν η πρώτη ωφελούμενη από αυτή την ε, ιδέα της ποσόστοσης, εγώ είμαι κατά της ε, πρότασης αυτής. Έχουμε λοιπόν πολύ καλές εξελίξεις. Είμαστε σχεδόν ευτυχείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το μόνο που μας έλειπε ακόμα θα ήταν να υπάρχει μια σαφής δομή που μας έχουν υποσχεθεί στην τελευταία ανάλυση για τη διαχείριση των κρίσεων και την πρόληψη των συγκρούσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πιοτρόφσκι για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, ευχαριστώ πολύ. Με λύπη μας διαπιστώνουμε πως μέλη της Επιτροπής των Εξωτερικών ε, ζητούν ε, ε, με σαν πρώτο αίτημα την γεωγραφική ε, κατανομή των μελών του προσωπικού της υπηρεσίας αυτής και το αίτημά τους απορρίπτεται. Οι ιδέες της ανταγωνιστικότητας, της ισότιμης ε, μεταχείρισης δεν μπορούν να επισκεφτούν από τις φιλοδοξίες των μεγάλων κρατών. Πρέπει όλοι να βρουν τη θέση τους σε αυτή την υπηρεσία η κυρία Άρστον έχει διακριτική ευχέρεια προς την υπόθεση των επιλογών για τις 150 θέσεων ε, ε, της υπηρεσίας της και βλέπουμε ότι σε σχέση με την Πολωνία που είναι σε ε, εξαπλάσια σε μέγεθος εμείς έχουμε μόνο δύο θέσεις Πώς αποφασίζεται λοιπόν αυτό το κοινοβούλιο, αποφασίζει μόνο τον προπολογισμό αυτή τη νέα διπλωματική αρχή που θα δημιουργηθεί. Ο Μπαλτασάρα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά από την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου για την ΕΕΔ, εμείς ε, σήμερα θέλουμε να καταστήσουμε λιταργική αυτή την απόφαση μέσα από τη χρηματοδότηση του της υπηρεσίας και το καταστατικό των υπαλλήλων. Θέλω να σταθώ σε μία πτυχή αυτής ε, της ε, έκθεσης που αφορά στη σύνθεση του προσωπικού, του διπλωματικού προσωπικού της υπηρεσίας. Άλλοι θα θέλανε μια διαφορετική ε, επιλογή του προσωπικού βασισμένη στη γεωγραφική προέλευση και στο φύλλο. Ευτυχώς καταφέραμε εμείς να περάσουμε αυτό το κριτήριο χωρίς όμως να επιβάλλουμε ποσοστώσεις εθνικού χαρακτήρα γιατί αυτό δεν θα ήταν καθόλου καλό. Μετά από 50 χρόνια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δημιουργείται σήμερα η πραγματική διπλωματική υπηρεσία της Ένωσης η οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει μια κοινή εξωτερική πολιτική και να θέσει ε, στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές τις υπηρεσίες. Πρέπει να συμμετέχουν σε αυτήν την υπηρεσία οι υπάλληλοι βάσει των κριτηρίων που εγκρίναμε στη νομική υπηρεσία εγκρίνοντας την έκθεση ΡΑΠΚΑΙ και διακόπτη πρόεδρος. Ευχαριστώ ο κύριος Τάλερ, να πάμε ομολητής παρακαλώ για ένα λεπτό. Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση 27 κρατών μελών και όχι μια ε, μειοψηφία. Ευχόμεθα κάθε επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, Υπηρεσία Εξωτερικής δράση. Τη χρειάζονται οι πολίτες, οι λαοί. Αλλά πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία αυτή ε, θα ε, υιοθετηθεί από όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα είναι επιτυχής, ότι θα είναι η ελίτ, η κρέμ, το της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη να εμπλακούν. Δεν μπορούμε ε, να ε, θέσουμε σε κίνδυνο την υπηρεσία αυτή με έξι εθνικότητες που να εκπροσωπούνται, έξι κρατημέλη που να εκπροσωπούνται ε, στην, στα νότερα στελέχη της υπηρεσίας. Τι γίνεται με τα άλλα κρατημέλη, με τα νέα κρατημέλη. Ελπίζω ότι δεν θα αγνοήσετε τις αποφάσεις του, των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω ότι τουλάχιστον σε 10 χρόνια θα έχει διορθωθεί η κατάσταση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σίβιτς για ένα λεπτό επίσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ολοκληρώνουμε πλέον μια νέα διαδικασία με μια νέα υπηρεσία και εγώ που εκπροσωπώ την Πολωνία, νέο κράτος μέλος, ε, παρασύρομαι από τον ενθουσιασμό όταν βλέπω ότι βρισκόμαστε πια στην ίδια την καρδιά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όταν βλέπουμε ότι αυτή η υπηρεσία είναι ο καρπός μιας συνεργασίας μεταξύ των οργάνων. Ε, το Κοινοβούλιο, ε, ε, ήταν ιδιαίτερα ενεργό βέβαια στην υπόθεση αυτή. Το μωρό αυτό λοιπόν είναι κοινό πεδίο όλων των θεσμικών οργάνων και ουσιαστικά έκφραση της συνεργασίας μεταξύ παλαιών κρατών μελών. Μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι λαμπρό, μπορεί να μην είναι δέκα με τόνο, αλλά ένα 9, μισή ίσως. Κυρία Άστον, εσείς με πολύ διαφανείς αποφάσεις που χρειάζονται αποφάσεις περί αξιοκρατικής επιλογής μπορείτε να κερδίσετε τις εντυπώσεις. Εάν δούμε ότι επιλέγετε κανείς με, τις, ε, με την αξία του και όχι για άλλους λόγους, τότε θα σας στηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φλάσσονο, κυρία Μπένοβα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συναδελφοί, κυρία Άστον, κύριε Επίτροπε, μιλάμε για μια μοναδική στιγμή σήμερα τη στιγμή της ίδρυσης της εξωτερικής υπηρεσίας, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ναι, μπορεί ο καθένα να έχει τις ε, κόκκινες γραμμές του, όμως βλέπουμε ότι μπόρεσαν οι συγγητέ να επεξεργαστούν μία ε, έκθεση αποδεκτή για τους πάντες. Ελπίζω αύριο το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει αυτή τη συμβαστική λύση. Με λύπη μου βλέπω ότι πολλοί από τους ε, εισηγητέ αναφερόμενοι στο θέμα αυτό περιορίστηκαν μόνο σε μία πτυχή, δηλαδή τη γεωγραφική εκπροσώπηση του προσωπικού. Η ιδέα, το μέλλον, το όραμα αυτής της υπηρεσίας δεν αναφέρθηκε παρκώς. Μα εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία της προσπάθειάς μας. Αυτή η διπλωματική υπηρεσία μπορεί να ξανακερδίσει την Ευρώπη μπορεί να την ξανακάνει μεγάλη δύναμη στην παγκόσμια σκηνή. Και πιστεύω κυρία Άρστον, ότι θα επιλέξετε μία ομάδα συνεργατών που θα εκπροσωπεί όχι μόνο τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πάνω απ' όλα θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως όλων, ως κοινό εγχείρημα όλων μας. Ευχαριστώ πολύ και τώρα περνάμε στη διαδικασία του ΚΑΤΣΤΙΑΕ. Και πάλι θα δώσουμε το λόγο ως ήθιστες, ε, όσο δυνατόν περισσότερους συναδέλφους, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος λοιπόν και για αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαι αυστηρή ως προς τον χρόνο ομιλίας. Η κυρία Κώστιγκερ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα διαδραματίσει από εδώ και μπρος την ε, το πιο σημαντικό ρόλο στην εξωτερική ε, εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εκπροσώπηση της στην παγκόσμια σκηνή και γι' αυτό θέλουμε να είναι στο δυνατόν πιο ε, επικοδομητική και απρόσκοπτη εργασία της. Ιδιαίτερα ή το θέμα της διαφύλαξης των δημοσιονομικών, της ομαλής λειτουργίας των δημοσιονομικών, όπως καταγράφεται στις εκθέσεις ε, Γκρέσλι και Ριμπελίνη, θα ήθελα να δοθεί έμφαση. Ιδιαίτερα δε με τις δηλώσεις αξιοπιστίας που κατατίθεται κάθε χρόνο, με τις εκθέσεις που θα είναι αναλυτικές θα υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο και την ε, έκθεση απαλλαγής που θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο για τον προπολογισμό της υπηρεσίας αυτής. Η έκθεση λοιπόν που έχει κατευθεί για μένα είναι πολύ καλή, αποτελεί το σωστό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Χάουιτ. Πρόεδρε, θα ήθελα ξεκινώντας να συγχαρώ την ύπατη εκπρόσωπο η οποία κατάφερε σήμερα να αλλάξει έδρανο στο Κοινοβούλιο, πέρασε από τη μία μεριά του Κοινοβουλίου στην άλλη, από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Συνήθως όποιος το κάνει αυτό χάνει και από αξιοπιστία και από υποστήριξη. Ε, ίσως κάποιοι συνάδελφοι θελήσουν να κάτσουν με το χρονόμετρο και να δουν πόση ώρα μείνατε στα έδρανα τη Επιτροπή και πόσα στα έδρανα του Συμβουλίου. Αλλά πάντω εύχομαι να έχετε πολύ καλή επιτυχία στη δουλειά σας και να, θα ήθελα να πω ότι ελπίζω να είναι αυτή η υπηρεσία ακριβώς αυτό το οποίο προβλέπει η συνθήκη να εκφράζει τα συμφέροντα, τα κοινά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να στρατευτείτε κι εσείς για μια πολύ καλή, αποτελεσματική και αντιπροσωπευτική υπηρεσία. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό και στο, στο έργο σας και γι' αυτό θα σας περιψηφίσω αύριο. Ευχαριστώ πολύ κύριος Βάγκελ, έχει το λόγο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, και μέλη το να βρεθούν συμβιβασμοί για τα οικονομικά αυτής της υπηρεσίας ήταν τόσο περίπλοκο θέμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονίσουμε τα συμφέροντά μας, διότι έχουμε διαφορετική ιστορία αλλά νομίζω ότι ο κοινό νους, η καλή θέληση και η προθυμία έχουν ίση κατανομή στην Ευρώπη και αυτό μας επιτρέπει να ε, διανοίξουμε ένα μέλλον ε, για την Ευρώπη. Στο μέλλον η εξωτερική πολιτική και ο ρόλος της Ευρώπης ε, σε διεθνές επίπεδο θα είναι στο επίκεντρο όπως τώρα Ε, οικονομικές ε, τα οικονομικά θέματα είναι στο επίκεντρο. Η Λέιδη Άστον και άλλοι θα διαμορφώσουν αυτή την πολιτική και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται πολύ για το θέμα αυτό. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ, πολύ. Επανέλθω στο θέμα της αξίας. Μια προστιθέμενη αξία που πρέπει να επιτευχθεί είναι στην συνεκτική πολιτική για την ανάπτυξη. Έχετε δεσμευθεί γι' αυτό. Πρέπει την προτεραιότητα αυτή να αντανακλάται στην πολιτική του προσωπικού, στην εκπαίδευση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόληψη των συγκρούσεων ε, αυτές οι δεσμεύσεις πρέπει να υπάρχουν ακόμα και στην εκπαίδευση και αυτό θέλουμε να δούμε από την 1η Δεκεμβρίου και μετά. Ευχαριστώ Πάσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης βραδύτατα αναπτύσσει τις δραστηριότητες της. Σήμερα συζητούμε την χρηματοδότηση της υπηρεσίας. Σχετικά με το θέμα αυτό, λέει Διάστον, πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι οι πόροι για την χρηματοδότηση όλων των θεσμικών οργάνων προέρχονται από τα κράτη-μέλη και η υπηρεσία αυτή στο τέλος θα ζήσει από τα χρήματα που θα προέρχονται από 27 κράτη-μέλη. Πρέπει να τα κατανοήσετε αυτό, κυρία Άστον. Ακόμη και αν συζητούμε για τα προσόντα για την επιλογή των διπλωματών, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ισορροπία τη γεωγραφική. Διότι το να μην εκπροσωπείται κανείς στα υψηλά επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να προκαλέσει ένα συνέστημα ότι ορισμένα ε, κράτη-μέλη δεν την χάνουν του δέοντος σεβασμού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε ότι η ΕΕΔ είναι μια ιστορική ευκαιρία για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Αλλά αυτό όμως έχοντας και μεγάλα οράματα διότι δεν είναι η ώρα τώρα για εσωτερικές διαμάχες ε, γύρω από τα κονδύλια και πολέμους μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε σήμερα είναι να έχουμε ένα γενικότερο όραμα για το πώς πρέπει να είναι η Ευρώπη ανά τον κόσμο. Το αντίθετο δηλαδή από αυτό το οποίο συνέβη μέχρι σήμερα. Όπως έγινε δηλαδή με το ε, με τον Νόμπελ, με Ειρήνης όπου ο καθένας είπε το κοντό του και το μακρύ του για αυτό το βραβείο. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να είμαστε ενωμένοι και να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Προέδρου μας του κυρίου Μπούζεκ. Ευχαριστώ πολύ. Συλλοφληρώθηκε η διαδικασία Κατστιάη και τώρα περνούμε στις δευτερολογίες. Η κυρία Άστον παρακαλώ. Έχει το λόγο. Πρόεδρε, πολύ σύντομα και από την άλλη πλευρά της Ολομέλειας. Ελπίζω να έκαθασα αρκετά λεπτά από τη μια και από την άλλη πλευρά. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τις παρεμβάσεις των, βουλευτές, των βουλευτών. Ιδιαίτερα καταγραφώ τις, ε, την επιθυμία γεωγραφική εκπροσώπηση και αξιοκρατία. Ιδιαίτερα καταγράφω την ε, δομή για τη διαχείριση των κρίσεων μέσα στην υπηρεσία. Ιδιαίτερα καταγράφω την ε, ενσωμάτωση της αρχής ε, των ανθρωπινών δικαιωμάτων σε κάθε δράση της υπηρεσίας μας και ιδιαίτερα καταγράφω τις δημοσιονομικές αρχές και την εκτέλεση του προπολογισμού. Και το ότι οι βουλευτές θέλουν μια αποτελεσματική υπηρεσία που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά και οικονομικά τα κονδύλια του προπολογισμού τη. Και ύστερα από όλου αυτού του μήνε των πραγματεύσεων καταγράφω τη βούληση του Κοινοβουλίου για μια υπηρεσία που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των ε, πολιτών της Ευρώπης που θα εκπροσωπεί καλά την Ευρώπη στην εξωτερική σκηνή. Όλα αυτά τα καταγράφω και ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και τώρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Επίτροπη, ο κύριο Λεβαντόφσκι, ο κύριο Σεφσκοβιτ, μετά και παρακαλώ όσο το δυνατόν πιο σύντομα γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Κύριε Λεβαντόφσκι, κύριε Πρόεδρε, πολύ πολύ σύντομα μια απάντηση στην κυρία Αντρίσεν που έχει ήδη αποχωρήσει για το ζήτημα της ουδετερότητας τη μοσονομικής υπηρεσία. Εμείς πιστεύουμε ότι μακροπρόθεσμα και με την εξοικονόμηση πόρων από τις ε, εθνικές δημοκρατικές υπηρεσίες και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η υπηρεσία εξωτερική δράση θα αποδείξει ότι είναι ε, δημοσιονομικά ουδέτερα. Ήταν λοιπόν προ το παρόν αυτή η λύση ε, μόνο κατάλληλη και αρμόσια και γι' αυτό υπόθηκε ότι θα πρέπει το 2013 να επανεξεργαστούν όλα αυτά με την μεσοπρόθεσμη ε, αναθεώρηση. Και κατά τα άλλα, άλλα σχόλια δεν θα κάνω. Αναμονή τη αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Σεύτσοβιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη για την υποστήριξα και την θετική ατμόσφαιρα της συζήτησης αυτής και επίσης συγχαίρουμε και το Συμβούλιο για την σημαντική συμβολή τους όλη αυτή την άσκηση και αυτή η θετική ατμόσφαιρα ε, μας έφερε κοντά στην ιστορική απόφαση που θα ληφθεί αύριο. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στους ευρωβουλευτές που μπόρεσαν να καταστήσουν εφικτή αυτή τη θετική ατμόσφαιρα και θα ήθελα να ευχηθώ κάθε τύχη στη νέα υπηρεσία και στην επικεφαλής ε, που θα έχει μια συνεκτική και συντονισμένη εξωτερική πολιτική διότι είμαι βέβαιος, είμαι πεπισμένο ότι με την πάροδο των ετών η Ευρώπη θα αυξήσει την παρουσία της ε, και τον ρόλο τη ε, στι διεθνείς υποθέσεις. Ελπίζω ότι θα έχουμε στενή συνεργασία και συνέργειε μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για ιδιαίτερα για τις σύντομες απαντήσεις που μας δώσατε. Μας βοηθάτε να τηρήσουμε το χρονοδιαγραμμά μας. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Ράπκα, ο συζητητής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ύστερα από τις ε, εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις, κατά την έναρξη της συζήτησης, έχω μόνο δύο παρατηρήσεις να κάνω. Ήθελα μάλιστα να το κάνω ούτως ή άλλως στο τέλος της συζήτησης, να ευχαριστήσω όλες και όλους τους κοιόδης συγητές. Αυτό βέβαια αποτελεί βασική προϋπόθεση της ε, κοινοβουλευτικής δουλειάς, αλλά ταυτόχρονα βοηθάει και τον εισηγητή όταν ξέρει ότι οι σκιώδεις εισηγητές είναι στο πλευρό του. Πρώτη παρατήρηση, γιατί οι διαπραγματεύσει δεν ήταν καθόλου εύκολε. Και δεύτερον, το ζήτημα του, της γεωγραφικής εκπροσώπησης. Η κυρία Νάινσκι είπε ότι δεν προβλέπεται τίποτα στον συμβασμό. Θα σας πω το εξής. Εφόσον τώρα έχουμε συμφωνήσει και πλέον μπορούμε να κάτσουμε με την ησυχία μας να διαβάσουμε τα κείμενα. Να διαβάσουμε τα κείμενα, να διαβάσουμε τα κείμενα γιατί όποιος διαβάζει τα κείμενα βλέπει και ενημερώνεται και καταλαβαίνει ότι υπάρχουν και δεσμευτικές ακόμη διατάξεις για τη γεωγραφική εκπροσώπηση και έτσι μπορείτε να σας καθασυχάσω. Ευχαριστώ πολύ και για άλλη μια φορά το λόγο θα λάβει τώρα ο κύριος Γουαλτιέρη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, Βεβαίως είμαι πολύ ικανοποιημένος για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι η εργασία που είχαμε ήταν δύσκολη αλλά πάρα πολύ σημαντική διότι να ενοποιήσουμε τις λειτουργίες που συνδέονται με διαφορετικές πολιτικές και διαδικασίες για να ενισχύσουμε την συνεκτικότητα της εξωτερικής δράσης Ένωσης χωρίς να κινδυνεύσει ο κοινοτικός χαρακτήρας ορισμένων πολιτικών αλλά ταυτόχρονα να ευνοήσουμε ορισμένες δομές για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας δεν ήταν απλώς διοικητικό θέμα γραφειοκρατικό θέμα, αλλά δοκιμασία των δυνάμεων ε, των οργάνων, αλλά έπρεπε να έχουμε ένα μέσο που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή και ε, να εξάρει και να αναβαθμίσει τον ρόλο της, ούτως ώστε να μπορεί η Ευρώπη ε, να δράσει περισσότερο στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στον Κάφκασο και στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι ότι αντιμετωπίσαμε αυτήν την πρόκληση. Μπορούμε λοιπόν να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι και η ύπατη εκπρόσωπος θα έχει την απαιτητική υποστήριξη αυτού του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε τη συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12.30. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές,